τη σύντομη παρουσία τη κυρία Φανμπόσοιτ, βελτίωσε τη νομοθεσία για την ενιαία αγορά. Το λόγο έχει η εισηγήτρια. Τέσσερα λεπτά. Ehm, Ευχαριστώ. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι ιδιαίτερως που επιτέλους έχω δυνατότητα να παρουσιάσω την έκθεσή μου για την βελτίωση νομοθεσία στην εσωτερική αγορά. Ήταν ένα μακρόπνοο σχέδιο και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα περνάει δύσκολους καιρούς με την ε, κρίση στην Ευρωζώνη, την κρίση του προσφυγικού, την κρίση στην ασφάλεια, τον Brexit, τον Grexit, το δημοψήφισμα στην Ολλανδία την περσμένη εβδομάδα και δεν μπορούμε πλέον να έχουμε τις παροπίδες. Πρέπει ε, να φύγουμε από αυτή την προσέγγιση ότι η περισσότερη Ευρώπη είναι η απάντηση σε όλα. Όταν με ρωτάει ο κόσμος τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για να προσελκύσει τα ενδιαφέρον των πολιτών της, η απάντηση που δίνω είναι ότι η Ευρώπη έχει η ίδια την ευθύνη να καταδείξει ότι ε, έχει κάποια ξένα προσδόση, ότι είναι σημαντική. Και μόνο τότε θα αναγνωρίσουν αυτή την αξία και οι πολίτες είναι και βεβαίως εν μέρη ευθύνη και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων με βάση βέβαια και την αρχή της επικουρικότητα, να καθορίσουν πότε θα πρέπει να αποφασίζεται κάτι ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή όχι, πότε θα πρέπει να παρεμβαίνουν ή όχι, με ποιον ε, τρόπο, αν απαραίτητη νομοθεσία και τελικά να φροντίζουμε και να μεριμνούμε ότι τα μέτρα ε, που υιοθετούμε θα είναι και εύκολα στην εφαρμογή τους. Και αυτή είναι και αφετηρία για την έκθεση για την καλύτερη νομοθεσία στην εσωτερική αγορά, που είναι ένα από του ακρογωνιαίου λήθου τη ευρωπαϊκή συνεργασία. Είναι πολύ σημαντικό η νομοθεσία που υιοθετείται και να μεταφέρεται στην εθνική νομοθεσία και να εφαρμόζεται από τα κρατή-μέλη. Ούτω ώστε να έχουμε απτά αποτελέσματα και να αντιμετωπίσουμε και τι προκλήσει τη ψηφιακή ενιαία αγορά ε, αλλά να έχουμε και τους ε, καρπούς που επιθυμούμε, πρέπει να λειτουργήσουν με αποφασιστικότητα τα θεσμικά όργανα. Ιδάλλως ε, μένουμε στάσιμοι. Με απλό και αποτελεσματικό τρόπο λοιπόν θα πρέπει να εφαρμόζουμε την νομοθεσία μας και διαρκώς να την αξιολογούμε ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι πάντα θα επιτυγχάνονται οι στόχοι μας. Η βελτίωση της νομοθεσίας ό,τι αφορά την ενιαία αγορά δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να καταργηθεί η νομοθεσία, η τμήμα της, όμως ότι θα πρέπει να έχουμε ένα ανταγωνιστικό κλίμα ως προς την νομοθεσία το οποίο θα διατηρήσει τις θέσεις εργασίας και τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Μια εσωτερική αγορά ε, που δίνει κίνητρα για την παραγωγή, την καινοτομία και το εμπόριο. Να τολμήσουμε λοιπόν να είμαστε και επικριτικοί και να θέτουμε ερωτήματα χωρίς ταμπού. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δώσουμε κίνητρα και δυναμική για την εσωτερική αγορά ε, και με μια μακροπρόθεσμη ανάπτυξη για την Ευρώπη και ευημερία για τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτή ήταν ε, η δική μου πρόταση και ελπίζω να τη στηρίξετε αύριο. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Διαδικασία Καριστιάη. Η κυρία Κοράτσα Πίλτ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαίρετη έκθεση. Καλύτερη νομοθεσία σημαίνει και καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Και αυτό δεν σημαίνει ούτε να περιορίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων και των καταναλωτών, αλλά, της γραφειοκρα... η γραφειοκρατία κυρίως. Πρέπει λοιπόν η ενιαία αγορά να παραμείνει απλή, αναλογική και εφαρμόσιμη στην ε, πραγματική οικονομία. Πρέπει να περάσουμε σε πραγματική ποιότητα και αξιολόγηση συνεπιών με μέτρα και εργαλεία όπως το Solvit που θα είναι στην υπηρεσία όλων των πολιτών. Ιδιαίτερα πρέπει οι εμπλεκόμενοι φορείς να συμμετέχουν στις διαδικασίες, πρέπει να αποφευθεί η περιττή επιβολή νομοθετικών ρυθμίσεων, ιδιαίτερα από τα κράτη-μέλη των εφαρμόζουν κανόνες εσωτερικής αγοράς και σε μια χρονική στιγμή όπου χρειάζεται διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στην ενιαία αγορά, που πρέπει να είμαστε πιο κοντά στο πολίτη, χρειάζεται υλοποίηση και όχι ιδεολογική αντιπαράθεση με τον πολίτη και τον καταναλωτή. Όπως είπε ο κύριος Τίμερμανς, ο αντιπρόεδρος, πρέπει να είμαστε μεγάλοι για τα μεγάλα θέματα και μικροί σε μικρή κλίματα, δηλαδή για τα μικρά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σάνι, ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία αυτή. Η εσωτερική αγορά έχει μεγάλη σημασία, η γενική αγορά έχει μεγάλη σημασία, η προστασία του καταναλωτή αποτελεί σημαντικό στοιχείο της. Ο καταναλωτή όμω. δεν ενημερώνεται πάντα, δεν είναι πάντα ενήμερο για τα δικαιώματά του και τον τρόπο να τα διεκδικήσει και να τα ασκήσει. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να προσφέρεται η πληροφόρηση στον καταναλωτή και να γίνεται η, ο συντονισμός με τις ενώσεις των καταναλωτών. Ένα σύστημα λοιπόν ε, κατάλληλο θα πρέπει να προσφέρει ένα πλαίσιο που θα παρακολουθεί την ε, τελευταία νομοθεσία, την καινοτομία ψηφιακή και, τεχνολογική, και άλλη τεχνολογική και πρέπει να σημειώσω εδώ ότι υπάρχει ε, μια τεχνολογία αιχμής ουγγρική η οποία σε επιτρέπει να διαβάζετε, επιτρέπει στα μηχανήματα να διαβάζουν το barcode ε, και τα σχετικά, σχετικές πληροφορίες. Ευχαριστώ κυρία Φόρτ για ένα λεπτό. Όχι. Η ενιαία αγορά στόχο έχει να διευκολύνει την επιχείρηση και τον καταναλωτή στις συναλλαγές τους μεταξύ 28 κρατών και 500 εκατομμύριων. Όχι επιπρόσθετο κόστος λοιπόν, αλλά λιγότερο κόστος πρέπει να φέρνει και να δημιουργεί έτσι θέσεις εργασίας, να εξασφαλίζει ανάπτυξη. Η έκθεση της Βελγίδας συναδέλφου που έχουν υποστηρίξει πολλοί σε άλλες χώρες σήμερα μας λέει ότι οι νέοι κανόνες πρέπει να εισάγονται όταν εξασφαλίζουν την ανάπτυξη των οικονομιών μας. Πρέπει να είναι απλοί και ε, ευχερεί στην εφαρμογή τους οι κανόνες, να είναι ε, μικρότερη επιβάρυνση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα εθνικά κοινοβούλια να έχουν ισχυρότερη φωνή και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη διαδικασία της κόκκινης κάρτας. Δεν είναι μόνη της λοιπόν η Βρετανία που ζητεί όταν ζητεί την ε, μεταρρύθμιση της Ευρώπης και χαίρομαι που μας υποστηρίζετε όλοι σήμερα. Ελπίζω αύριο στην Ολομέλεια να εγκριθεί από όλους τους συναδέλφους. Η έκθεση ευχαριστώ. Κύριος Καπούτο. you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το θέμα της ενιαίας αγοράς για να προωθήσουμε την ανάπτυξη και τις νέες θέσεις εργασίας αφορά ε, ένα πολύ σημαντικό μέρος αυτού του κόρπους έτσι ώστε να γίνουν ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις μας και έτσι ώστε να μας έχουν εμπιστοσύνη οι καταναλωτές. Μέσα στα πλαίσια της βελτιστοποίησης της αγοράς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την προστιθέμενη αξία της διακυβέρνησης και των ρυθμίσεων επικαιροποίησης. Πολλές φορές δεν υπάρχουν σωστοί δείκτες για να μπορέσουμε να μετρήσουμε την αποδοτικότητα της νομοθεσίας και πιστεύω ότι σε κάθε ε, κατεξιδότηση πράξη και εκτελεστική πράξη θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις βασικές αξίες που τις διέπουν, δηλαδή τη διαφάνεια και τη συνοχή. Κύριε Καπούτο, έχω εδώ μια κόκκινη λάμπα μπροστά μου ένα λαμπάκι κόκκινο, το οποίο ανάβει πάντα όταν ο ομιλητής είναι τόσο γρήγορος που δεν είναι σε θέση οι διερμηνείς να το μεταφράσουν. Ήταν αναμένο συνέχεια το λαμπάκι μου την ώρα που μιλούσατε. Και σας παρακαλώ πολύ για εκείνους συναδέλφους οι οποίοι δεν μπορούν να σας καταλάβουν στη γλώσσα σας να μιλάτε πιο αργά. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής παρακαλώ. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με την ε, έκθεση σε σχέση με την ε, καλώς ρυθμισμένη ενιαγορά. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει σωστή φιλοδοξία και η προστασία και η ασφάλεια ε, της κοινωνίας, καθώς και η καλύτερη εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου και να μην δημιουργήσουμε νέα όταν έχουμε την παλαιά που δεν, ε, την οποία δεν έχουμε χρησιμοποιήσει πλήρως για να υπάρξει μεγαλύτερη ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας και να βοηθήσουμε τις αναδυόμενες οικονομίες αλλά και τις επιχειρήσεις της ψηφιακής οικονομίας. Επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε τη μακροχρόνια ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ευημερία των πολιτών της. Ευχαριστώ τελευταία στο δικασία Καριστιά. Κυρία Τόμα λεπτό. Ευχαριστώ. Η ενιαία αγορά είναι υψή της σημασία εγχείρημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλέον ε, έχουμε συνηθίσει να υπάρχει ελεύθερο εμπόριο μεταξύ των χωρών μας και για να συνεχιστεί αυτή η ευημερία στην ενιαία αγορά θα πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις υπηρεσίες και να υπάρξει και προστασία απέναντι σε αθέμητες ε, πρακτικές ή εσφαλμένη εφαρμογή των ε, νομικών διατάξεων ή να, να προσπαθήσουμε τόσο ώστε να μην ζημιώνονται οι μικρές και μεσαίε επιχειρήσεις που αποτελούν και το 80% της εμπορικής δραστηριότητα. Πρέπει λοιπόν να περιορίσουμε το διοικητικό άχθος και να δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες στις μικρομεσαίε επιχειρήσεις. Αυτές θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητές μας. Ευχαριστώ πολύ. κύριε κυρία Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, Εξ ονόματο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ενία Αγορά και ιδίω ε, την εισηγήτρια κυρία Βαν Μπόσερτ για αυτή την έκθεση. Συμφωνούμε ότι η ενιαία αγορά αποτελεί ακραγωνιαίο λίθο τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Στι τελευταίε δεκαετίε έχει ε, δώσει περισσότερε θέσει απασχόληση και έχει συμβάλει ε, στην ανάπτυξη. Πρέπει λοιπόν να την εντάξουμε και να την εξετάσουμε από το πρίσμα του συνόλου του κύκλου πολιτικής. Πέρυσι λοιπόν εμείς παρουσιάσαμε δύο ε, πρωτοβουλίες, ε, την βελτίωση της νομοθεσίας και τη στρατηγική για την ενιαία αγορά. Τον περασμένο Μάιο, λοιπόν, προτείναμε το πακέτο για την βελτίωση τη νομοθεσία που καλύπτει ολόκληρο το κύκλο πολιτική, από τι αξιολογήσει μέχρι την υιοθέτηση, εφαρμογή και αξιολόγηση τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία το πακέτο αυτό θα μας ε, βοηθήσει να διασφαλίσουμε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία θα αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα των ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να βασιζόμαστε σε καλύτερα, πιο εύρωστα στοιχεία και πιο προσεκτική αξιολόγηση ε, του αντικτύπου. Αυτό θα μα επιτρέψει ε, να ανακτήσουμε και την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών. Και πρόσφατα είχαμε και μία διαπραγμάτευση ε, διοργανική για την βελτίωση της νομοθεσίας και πλέον έχουμε ένα πιο ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο και ανανεωμένη δέσμευση των επιμέρους θεσμικών οργάνων. Μετά την επίσημη υιοθέτησή του, θα πρέπει και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καλή εφαρμογή του πακέτου αυτού ούτω ώστε όλοι να βλέπουν ε, με πολύ απτό τρόπο και όχι μόνο θεωρητικά ε, τα πλεονεκτήματα αυτής της πολιτικής. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το δικό της ε, πρόγραμμα πιο συγκεκριμένα συμβάλλει σε αυτή την ε, προσπάθεια περικοπής ε, του περιτού διοικητικού άχθους, ιδίως ό,τι αφορά τις πολύ μικρές και τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Και αυτό θα το πράξουμε χωρίς να υποσκάψουμε τους ε, κοινωνικούς, εργασιακούς ή περιβαλλοντικούς μας σκοπούς. Η δεύτερη πρωτοβουλία που αναλάβαμε πέρυσι ήταν η στρατηγική για την ενιαία αγορά που υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο με τρεις βασικούς στόχους. Τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ενίσχυση της τις της εξυγχρονιστικής ε, που χρειάζεται η Ευρώπη και πάνω απ' όλα η διασφάλιση της ε, πρακτικής εφαρμογής με απτούς στόχους. με βασικούς ε, ε, κλάδους της οικονομίας, υιοθέτηση νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των διακρίσεων κατά των καταναλωτών, βάση της χώρας ε, διαμονής και με άλλους τρόπους. Όμως όλα αυτά δεν επαρκούν. Δεν φτάνει δηλαδή μόνο να έχουμε νέες πρωτοβουλίες, όμως πρέπει να μεριμνήσουμε και για την κατάλληλη και επαρκή εφαρμογή της νομοθεσίας, να έχουμε καλύτερο σχεδιασμό της νομοθεσίας και καλύτερη αξιολόγηση των όσων δεν πηγαίνουν όπως πρέπει. Και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι υφιστάμενοι κανόνες θα εφαρμόζονται με τον σωστό τρόπο από τα κράτη-μέλη και με μια ευφυή προσέγγιση για να αναπτύξουμε και μία κουλτούρα της συμμόρφωσης. Για παράδειγμα, θέλουμε μια βελτιωμένη και ενισχυμένη συνεργασία ε, και για την νέα νομοθεσία και ετήσιες ε, διαβουλεύσεις ως προς τη συμμόρφωση με όλα τα κράτη-μέλη. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, έχουμε τους ίδιους στόχους, το ίδιο ευρύ όραμα για τα όσα θέλουμε να πετύχουμε. Όλοι θέλουμε να βελτιώσουμε την νομοθεσία για την ενιαία αγορά και να έχουμε και καλύτερους στόχους, καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας. Ας εργαστούμε από κοινού λοιπόν για να το πετύχουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Επίτροπα.